Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 7 kwietnia 2011. Και για τη συνεδρίαση που είχε διακοπεί συνεχίζεται με τη σημερινή μας συνεδρία.